Uh, please take a standing position, colleagues. Will be European anthem. Παρακαλώ να μείνουμε όλοι όρθιοι για να ακούσουμε τον Ευρωπαϊκό ύμνο.

Αγαπητοί προσκεκλημένοι, κύριε Επίτροπε, κύριε Υπουργοί, είναι μεγάλη τιμή να σας παρουσιάσω την εξοχότητά του Αμαντού Τουρέ, πρόεδρο της Δημοκρατίας του Μαλή και τη σύζυγό του. Δεν έρχεται για πρώτη φορά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας του Μαλή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά είναι η πρώτη φορά όμως που θα ακούσουμε την ομιλία του. Μας είχε επισκεφθεί τον Απρίλιο του 2009, εδώ και 1,5 περίπου χρόνο. Η ομιλία του Πρόεδρου του Μαλή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, λίγο πριν από τη συνάντηση που θα οργανωθεί σε δύο εβδομάδες στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη σχετικά με τους στόχους της χιλιετίας. Ξέρουμε τα προβλήματα που αντιμετώπισε η χώρα τα τελευταίους μήνες και τον τελευταίο καιρό γενικότερα σε σχέση με την απειλή της τρομοκρατίας και πόσο εμπλέκεται στην προσπάθεια καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Η δημοκρατία του Μαλή είναι επίσης μία από τις χώρες της Αφρικής όπου ο εκδημοκρατισμός έχει κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου είναι ένα μεγάλο σημείο επιτυχίας θα έλεγα για την περιοχή αυτή της Αφρικής. Χάρη στον ηγετικό ρόλο του Προέδρου Τούρε, τα γεγονότα τα οποία εξελίχθηκαν από τις αρχές της δεκαετίας του 90 προχώρησαν σωστά μετά από δύο δεκαετίες στρατιωτικής εξουσίας οι αλλαγές προς τη δημοκρατία φαίνεται ότι βγάζουν πλέον ρίζες. Φυσικά υπάρχουν πολλά που μένει να γίνουν ακόμα. Είμαστε πάντα και είναι η χώρα αυτή σε διαδικασία μαθητείας. Παρ' όλα αυτά οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται, δεν έχουν διακοπή και υπάρχει ανάγκη λοιπόν και στη δημοκρατία του Μαλή να εμβαθυνθεί η δημοκρατία. Η παρουσία σας λοιπόν εδώ έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο ενημερωτικά για το τι συμβαίνει στην Αφρική και για το πώς η χώρα σας μπορεί να εκπροσωπεί το σύνολο της Αφρικανικής Υπήρου προς την δημοκρατική ανάπτυξη και την ελεύθερη οικονομία αλλά είναι σημαντικό και για μας εδώ το ότι βρίσκεται ανάμεσά μας, διότι θέλουμε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να είμαστε πρωτοπόροι στην βοήθεια που δίδεται προς τις χώρες αυτές, και θέλουμε να είμαστε επίσης πρωτοπόροι στην στήριξη των χωρών της Αφρικής που σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις βασικές αξίες τις οποίες ε, είναι εδρεωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι πεπισμένος λοιπόν ότι οι προσδοκίες και των δικών μας πολιτών είναι ταυτόσιμες με τις αντίστοιχες της Δημοκρατίας του Μαλή, των πολιτών της Δημοκρατίας του Μαλή και γι' αυτό με πάρα πολύ ενδιαφέρον περιμένω την ομιλία σας και σας δίδω αμέσως το λόγο. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριε Υπατή εκπρόσωπος για τα θέματα εξωτερικών υποθέσεων και την πολιτική ασφάλειας, κύριε Επίτροπε για την Ανάπτυξη, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές, αξιότιμοι βουλευτές του Μαλή. Καταρχήν θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να σας συγχαρώ για την εκλογή σας επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα όμως κυρίως να ευχαριστήσω θερμά τους Προέδρους των πολιτικών ομάδων και όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μου δίνουν το προνόμιο να είμαι σήμερα εδώ παρόν ώστε να μπορώ ε, να εκφράσω παρουσία σα ε, τι θέσει μου για κάποιες μεγάλες προκλήσει που αντιμετωπίζει η χώρα μου και ολόκληρη η Αφρική. Και ιδίως να επιμείνω στις προσπάθειες που καταβάλουμε καθημερινά, ούτω ώστε να βρεθεί η κατάλληλη λύση. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, το Μάλι έχει μια έκταση 1.240.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και βρίσκεται στο κέντρο της Δυτικής Αφρικής. Έχουμε 7 χώρες ε, γύρω-γύρω και 7.000 ε, χιλιόμετρα είναι το μήκος των συνόρων μας. Είναι μια χώρα με παλαιό πολιτισμό. Έχουμε μια πλούσια και πολυπίκυλη πολιτιστική κληρονομιά και η ιστορία του Μαλή είναι ιδιαίτερα πλούσια και θα μπορούσε κανείς να αναφέρει συγκεκριμένα συμβολικά γεγονότα. Θα ήθελα να αναφέρω τη χάρτα του Κούρουκαν Φουγκά που υιοθετήθηκε πριν από 776 χρόνια όταν ιδρύθηκε η αυτοκρατορία του Μάλι. Η χάρτα του Κουρουκάν Φουγκά ήταν αντίστοιχη ενός συντάγματος. Κωδικοποιούσε την οργάνωση των εξουσιών τους όρους, τους περιορισμούς, τις υποχρεώσεις, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ε, ε, δημόσιας της ελευθερίας των πολιτών και την διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών και, ε, των, και της περιουσίας τους. Το άτομο χέρι άκρας αξιοπρέπειας και δεν μπορούν να παραβιαστούν τα δικαιώματά του. Αυτά ήταν αυτά τα οποία θεσπίζει αυτός ο χάρτης και νομίζω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που πρεσβεύει αντίστοιχε αξίες. Η ιστορία του Μαλή είναι και το Τουμποκτού, η μυστηριώδης πόλη που ήδη από το 16ο αιώνα είχε 25.000 φοιτητές που είχαν έρθει από πολλές χώρες για να ακούσουν ε, τους σοφούς στο τζαμί του Σαν Κορέ και στο Πανεπιστήμιο γύρω από αυτό το τέμενος. Μαμού Καλκαντή μιλά για την εποχή αυτή και παραθέτω τα λόγια του. Το Τομπουκτού ήταν αναγνωρισμένο για το υψηλό επίπεδο των θεσμών του, για τις πολιτικές ελευθερίες, για τη διασφάλιση των ατόμων και των αγαθών τους, για την επίκαια προς τους φτωχούς και προς τους ξένους, για την ευγένεια προς τους φοιτητές και τους επιστήμονες και για τη βοήθεια που παρέχεται σε αυτούς τους φοιτητές και επιστήμονες. Το 2006 η πόλη του Τιμπουκτού ανακηρύχθηκε πρωτεύουσα του Ισλαμικού πολιτισμού. Το Μάλι είναι και η χώρα Ντογκόν, που είναι γνωστή για την ε, εξαιρετική γεωγραφική του θέση και για τον ε, πολιτιστικό του πλούτο και γι' αυτό είναι και μεγάλο το τουριστικό ρεύμα προς τη χώρα μας. Η ιστορία του Μάλι είναι η ιστορία των παλαιών σχέσεων που έχουμε με την Ευρώπη και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι ο πρέσβης Μασάν ε, Μουσά είχε διπλωματικές σχέσεις με την Πορτογαλία ήδη από το 14ο αιώνα. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές, ενώπιον σας, ενώπιον των εκλεγμένων εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη αναγνώριση του λαού του Μαλή για τη συνεργασία και την ποιότητα των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Σχέσεως και Δημοκρατίας του Μάλι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πρώτος εταίρος για την ανάπτυξη του Μαλή. Είμαστε ε, ο δεύτερος, ε, η δεύτερη χώρα που λαμβάνει κονδύλια για την ανάπτυξη στην Αφρική, νοτίως στη Σαχάρα. Θα ήθελα να σας διασφαλίσω, να σας διαβεβαιώσω για την καλή μας συνεργασία και θα ήθελα να αναφέρω ότι το ένα το πρόγραμμα για την ανάπτυξη υλοποιήθηκε κατά 100% και εδώ και δύο χρόνια περίπου εκτελείται και υλοποιείται με πολύ καλή, καλές βάσεις το επόμενο πρόγραμμα αναπτυξιακής ε, πολιτικής. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, ε, το αποτέλεσμα τη συνεργασία μα έχει άμεσε επιπτώσει στην ποιότητα ζωή του πληθυσμού. Παράλληλα, ενδυναμώνει και τη βάση του δημοκρατικού μα συστήματο. Μετά το ε, πραξικόπημα της 26ης Μαρτίου του 1991 υπήρξαν κάποια γεγονότα σταθμή στην ιστορία του Μαλή και σιγά σιγά φτάσαμε στην μετάβαση στη δημοκρατία στις 8 Ιουνίου του 1992 βάσει όλων των δεσμεύσεων που οφείλαμε να αναλάβουμε. Μέσα στους 14 αυτούς μήνες της μεταβατικής περίοδου οργανώθηκαν ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές το 1992 και 10 χρόνια αργότερα, το 2002, εξελέγην επικεφαλής μιας προεδρικής λίστας και εδώ έχουμε την πρώτη αναλογή εξουσίας με δημοκρατικό τρόπο στο Μαλί. Μετά, τις μετά την εκλογή μου, κυρίε και κύριοι, πρότεινα στους και στου πολιτικούς στη χώρα μου μέτρα τα οποία με δύο λόγια θα μπορούσα να τα εκφράσω ως εξής. Θα πρέπει να κυβερνήσουμε από κοινού και να σεβόμαστε τις διαφορές. Αυτή μας η προσπάθεια είναι μια συνειδητή προσπάθεια υπέρ της κοινωνικής πρόοδου και υπέρ της ανάπτυξης της δημοκρατίας του Μάλι. Η εξουσία, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να είναι ένας παράγον συνοχής και όχι ε, διαίρεσης. Παράλληλα τηρώντας όλα, όλες τις θεμελιώδεις ελευθερίας. Πρέπει να τονίσουμε ότι η πολιτική συνένεση την οποία ακολουθήσαμε και την οποία πρότεινα δεν σημαίνει ομοφωνία η συνένεση, σημαίνει ότι συμπεριλαμβάνεται η έννοια του συμβιβασμού. Η πολιτική συνένεση στο Μαλί είναι μια προηγμένη πρωτοβουλία προς την κατεύθυνση αυτού του νέου πολιτικού συστήματος το οποίο διαμορφώνεται σιγά σιγά στην Αφρική. Δηλαδή ένας ευρύς κυβερνητικός συνασπισμός. Οι προσδοκίες ε, στο Μαλί είναι να συνενωθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις γύρω από το όραμα ενός Προέδρου που θα είναι ανεξάρτητος ε, και εκλεγμένος. Αυτό θα αποτελέσει τη βάση της συμφιλίωσης μεταξύ όλων των συνιστοσών του πολιτικού φάσματος και μια συμφιλίωση μεταξύ όλων των πολιτικών των ιδίων. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές, μέσα σε αυτό το ίδιο πνεύμα συνένεσης, ακολούθησε ο προβληματισμός μας για την παγίωση της δημοκρατίας στο Μαλί, μετά από 20 χρόνια άσκησης της εξουσίας. Η Επιτροπή που είναι υπεύθυνη για αυτό το έργο συναντήθηκε με όλους τους πολιτικούς ηθήνοντες, με την κοινωνία των πολιτών, με τους εκπροσώπους ε, των θρησκειών, ε, με τα συνδικάτα και με όλους τους ε, νομιμοποιημένους φορείς και από αυτή τη διαβούλευση ο στόχος μας είναι να διορθώσουμε τα κενά και τις ανεπάρκειες που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια άσκησης του θεσμικού έργου. Θέλουμε να έχουμε μία ισχυρή συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές και να μειώσουμε το κόστος των εκλογικών αναμετρήσεων. Θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα καταστατικό και για την αντιπολίτευση και για τους επικεφαλείς της αντιπολίτευσης. Όλα αυτά θα είναι αντικείμενο ενός συνταγματικού δημοψηφίσματος μετά την έγκρισή τους από την Εθνική Συνέλευση του Μαλή. Εδώ θα ήθελα ενώπιόν σας να αποτείνω ένα φόρο τιμή προς τους βουλευτές του Μαλή, με τους οποίους έχω άριστες σχέσεις. Και με τους βουλευτές της προεδρικής πλειοψηφίας και με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Και θα ήθελα να εκφράσω προς όλους τους βουλευτές του Μαλή τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες, διότι δέχθηκαν να με συνοδεύσουν εδώ και να είναι παρόντες σήμερα εδώ στο Στρασβούργο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριε και κύριοι βουλευτέ, η πολιτική και θεσμική εξέλιξη του Μαλή πάντοτε θα αφήνει ιδιαίτερο χώρο για την αποκέντρωση και θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι είμαστε μια μεγάλη αυτοκρατορία και γνωρίσαμε ε, πολλά στην ιστορία μας. Από το 13ο αιώνα η αποκέντρωση ήταν κάτι το οποίο το εφαρμόσαμε στην πράξη. Και οι περιφερειακές προσεγγίσεις για την αποκέντρωση βασίζονται στους εξής παράγοντες. Καταρχήν υπάρχει η πολιτική βάση εναρμονισμένη με την πεποίθηση ότι η αποκέντρωση δεν μπορεί να επιτύχει χωρίς την ανάθεση σταδιακά στις περιφερειακές αρχές όλων των καθηκόντων. Δεν μπορεί να επιτύχει χωρίς τη διαμόρφωση και εφαρμογή των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων για να βελτιωθεί η οικονομική και κοινωνική διακυβέρνηση και κυρίως σε τοπικό επίπεδο. Δεν μπορεί να επιτύχει χωρίς την επιδίωξη και ε, την παρακολούθηση ε, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από πλευράς χρηματοδότησης και από πλευράς ε, τεχνικής. Υπάρχει τρίξης διοικητικών μεταρρυθμίσεων που επωφελήθηκαν από την στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οδηγούν σε καλύτερη οργάνωση του κράτους και εξυγχρονισμό της διοίκησης, ενισχύοντας τις δυνατότητες ε, του κράτους. Έχουμε ε, 703 ε, περιφέρειες ε, και 49 ε, κοινότητες που είναι αντικείμενο διαχείρισης από περιφερειακά και τοπικά συμβούλια και υπάρχει ένα μεγάλο περιφερειακό συμβούλιο που διασφαλίζει την εκπροσώπηση όλων αυτών των οντοτήτων κατά τρόπο αποκεντρωμένο. Η δημιουργία μια γερουσία επίση είναι κάτι το οποίο έχουμε κατά νου στι πολιτικέ μεταρρυθμίσει που προτείνονται για να εμβαθύνουμε τη διαδικασία αποκέντρωση. Για να στηρίξουμε την τοπική ανάπτυξη, έχουμε επιλέξει ένα πρωτότυπο χρηματοδοτικό όργανο, που είναι ο Εθνικός Φορέας Τοπικών ε, Οντοτήτων και έχει επιτρέψει να υλοποιηθούν πολλές τοπικές επενδύσεις και να προσφέρονται βασικές κοινωνικές υπηρεσίες στον πληθυσμό του Μαλή. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι βουλευτές, Ενώπιον ε, της ε, Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ήθελα να δείξω και το θέμα της μετανάστευσης. Το θέμα της μετανάστευσης μας αγγίζει όλους, διότι για καθέναν από εμά, για κάθε χώρα, έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα. Και μέσα στον ίδιο προβληματισμό εντάσσονται και δημογραφικά θέματα και οικονομικά θέματα και κοινωνικά θέματα ανθρωπιστικά, καθώς και θέματα ταυτότητας και θέματα ασφάλειας. Σήμερα πρέπει να βρούμε κοινού ε, ε, τόπους ε, συζήτησης και κοινά συμφέροντα, ούτως ώστε η μετανάστευση να είναι ένας παράγων που θα συνεισφέρει στη συνολική ανάπτυξη και των δύο υπήρων μας. Αυτή είναι η πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε. Η διαρροή εγκεφάλων αποτελεί το πιο σημαντικό κόστος της μετανάστευσης για τις αφρικανικές χώρες. Λαμβάνοντας υπόψη το μικρό αριθμό εξειδικευμένων στελεχών και στην εκπαίδευση και στην υγεία. Σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, 40% των αφρικανικών χωρών Ε, ε, έχουν το 35% των πτυχιούχων τους ε, να διαμένουν στο εξωτερικό. Η μετανάστευση όμως στην Αφρική είναι μετανάστευση που διεξάγεται στην Αφρική. Από το 1 δισεκατομμύριο Αφρικανών που θεωρούνται μετανάστες, μόνο 2 εκατομμύρια θεωρείται ότι ζουν στην Ευρώπη από τους Αφρικανούς κάτω τη Σαχάρα όλοι αυτοί, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, διασχίζουν την έρημο, τη θάλασσα, τους ωκεανούς για να φτάσουν την Ευρωπαϊκή Ήπειρο εν είδη παραδείσου. από αυτούς σκεφτείτε πόσοι έχουν πεθάνει από δίψα ή πόσοι έχουν πνιγεί διασχίζοντας τη θάλασσα. Δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν στατιστικά δεδομένα για να μας δώσουν τέτοιο αποτέλεσμα. Και θα σας δώσω το παράδειγμα της χώρας μου. Η Δημοκρατία του Μάλι, που είναι μια μεγάλη χώρα μετανάστευση από και προς το Μαλί από τα 4 εκατομμύρια των κατοίκων του Μαλή που βρίσκονται σε ολόκληρο τον κόσμο, τα 3,5 εκατομμύρια ζουν στην Αφρικανική Ήπειρο και περίπου 200.000 σε ολόκληρη την Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Από οικονομικής απόψεως, η μεταφορά εισοδημάτων της διασποράς υπολογίζεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, το 1% του ΑΕΠ, σύμφωνα με μια μελέτη της Αφρικανικής Τράπεζας Ανάπτυξης που έγινε το 2005. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, αυτή η μεταφορά εμβασμάτων από τη διασπορά αντιστοιχεί στο 85% της αναπτυξιακής βοήθειας που δίδεται στο Μαλί. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να χαιρετήσω την ποιότητα του πολιτικού διαλόγου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαλή για τα θέματα της μετανάστευσης. Η ανάπτυξη είναι κάτι το κεκτημένο και δίνει τη δυνατότητα στους εταίρους μας να χρηματοδοτήσουν προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης των νέων σε διάφορα επαγγέλματα και να υποστηρίξουν πρωτοβουλίες για τοπική απασχολησιμότητα και ανάπτυξη της των ε, δεξιοτήτων επιτόπου. μα δόθηκε η δυνατότητα να ξεκινήσουμε και μια πιλωτική εμπειρία δημιουργώντας ε, το Κέντρο πληροφόρηση και Διαχείρισης μετανάστευση στον Παμάκο και η αποστολή αυτού του κέντρου είναι η βελτίωση των γνώσεων σχετικά με το φαινόμενο της μετανάστευσης καθώς ε, και η παροχή κατευθυντήριων ε, γραμμών και η, παρακολούθηση και η συνοδεία προς τους ε, προερχόμενους από το Μαλί για την επάνωδο στη χώρα τους. Θέλουμε να ευαισθητοποιήσουμε τον πληθυσμό για να αποφεύγεται η παράνομη μετανάστευση. Ακόμη θέλουμε να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο κεφάλαιο και από οικονομικής και από τεχνικής πλευράς όπως εκπροσωπείται από τους πολίτες του Μαλή που ζουν στο εξωτερικό. Το θέμα της ασφάλειας αποτελεί μια σημαντική πτυχή των ανταλλαγών μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό είναι σκόπιμο να ασχοληθείτε με το θέμα ε, του Σαχέλ ε, που είναι σημαντικό και για την Ευρώπη. 8 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα καλύπτονται, το 1 τέταρτο δηλαδή ε, της Αφρικανικής Επίρου και εκτείνεται από τη Μαυριτανία μέχρι το Σουδάν. Και καλύπτεται και το Μαλί και η Μπουρκίνα Φάσο και ο Νίγηρας και η Αλγερία και η Λιβύη και το Τσάντ. Η περιοχή Σαχάρα Σαέλ έχει σχεδόν μηδενική πυκνότητα ε, κατοίκησης. Είναι ένας ορεινός όγκος ε, επί, πολλά, ε, επί εκατοντάδες χιλιόμετρα και παράλληλα αμόλοφοι, γεωγραφικές συνθήκες δηλαδή, ιδιαίτερα αντίξωες, η θερμοκρασία μπορεί να είναι ένας βαθμός το Δεκέμβριο και από το Φεβρουάριο και μετά μπορεί να είναι 50 βαθμοί υποσκιάν. Η εντατική γεωργία είναι η μοναδική δραστηριότητα σε ένα περιβάλλον καθόλου φιλόξενο. Φέτος χάσαμε περίπου το 50% του αριθμού των ζώων στην ζώνη της Σαχάρας. Οι πληθυσμοί ε, ζουν πάρα πολύ δύσκολα και η νεότητα δεν έχει καμία άλλη εναλλακτική λύση από το να προσφεύγει σε εγκληματικές δραστηριότητες που ελέγχονται από άλλους κύκλους και αυτό είναι ένας μόνιμος κίνδυνος για τη χώρα μου το Μαλί το οποίο βρίσκεται στην κεντρική δυτική πλευρά καλύπτει περίπου 500.000 τετραγωνικά μέτρα, 70 περίπου της 100 δηλαδή του συνόλου της χώρας ανήκει στη Σαχάρα. Είναι μια χώρα διαμετακόμισης επίσης, είναι μια χώρα όμοιρος και θύμα κάποιων μεθοριακών απειλών οι οποίες προέρχονται από συγκρούσεις οι οποίες δεν είναι τοπικές αλλά ανήκουν σε άλλες χώρες. Υπάρχει λαθρεμπόριο, υπάρχουν ναρκωτικά, υπάρχουν ελαθρέα τσιγάρα, υπάρχει φυσικά και έλεγχος της παράνομης μετανάστευσης και υπάρχουν και οι λεγόμενες ομάδες των φανατικών Ισλαμιστών, οι σαλαφιστές τα χαρακτηριστικά όλων αυτών των παράνομων δραστηριοτήτων ε, οδηγούν θα έλεγα στο να είναι η περιοχή μας ιδιαίτερα εύθραυστη. Καμία από τις απειλές αυτές ε, οι τις οποίες προανέφερα δεν γεννήθηκε στο Μαλί. Καμία από τις ε, απειλές αυτές δεν ανήκει στη χώρα μου. Η χώρα μου είναι μια χώρα χωρίς επίσημο θρήσκευμα. Φυσικά το Ισλάμ ε, υπάρχει στη χώρα μου από τον 16ο αιώνα αλλά πάντα το Ισλάμ ε, το πιστεύει ο κόσμος στο Μαλί με ειρηνικό τρόπο και είναι απαράδεκτο το να προωθούνται ιδεολογίες Ισλαμιστικές στη ζώνη αυτή της Σαχάρας. είναι εντελώς ακατανόητη η ιδεολογία του πολιτικού Ισλάμ για μας. Οι επιπτώσεις οι θρησκευτικές που έχει αυτή η ιδεολογία είναι απαράδεκτες και για πόσο καιρό θα υφιστάμεθα τέτοιες απειλές. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Κυρίες και κύριοι, οι χώρες της περιοχής αυτής της υποσαχαρικής Αφρικής, ιδιαίτερα και του Μαλή, κάνουν τεράστιες προσπάθειες και σε ανθρώπινο επίπεδο και σε οικονομικό επίπεδο για να αντιμετωπίσουν τον διαμεθοριακό χαρακτήρα της ανασφάλειας η οποία αυξάνεται συνεχώς. Η ευρύτητα αυτού του φαινομένου νομίζω ότι τεκμηριώνει την υιοθέτηση από πλευράς του Μαλή μιας εθνικής πολιτικής ασφαλείας, καταπολέμηση μάλλον της τρομοκρατίας στην περιοχή αυτή της σαχάρα. Η πολιτική αυτή θα βασίζεται κυρίω στην σωστή πλαισίωση και φύλαξη των πληθυσμών έτσι ώστε να εφαρμοστούν σωστά οι πολιτικές ασφάλειας, στην βοήθεια στις εύθραυστες κατηγορίες του πληθυσμού καλύπτοντας τις βασικές τους ανάγκες και επίσης στην παροχή των βασικών κοινωνικών υπηρεσιών. Για να εφαρμοστούν όλα αυτές οι πολιτικές λοιπόν πρέπει ε, να ενισχυθεί το πρόγραμμα συλλογής όλων των μικρών όπλων το οποίο έχει ξεκινήσει όπως επίσης και η βελτίωση μιας περιφερειακής ή καλύτερα υποπεριφερειακής συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες έτσι ώστε να μπορέσουμε να δείξουμε πόσο βάρος δίδουμε στην προσπάθειά μας. Το Μαλί ε, έχει κάνει προτάσεις και αναλύσεις ε, για, τις, ε, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Οι αναλύσεις αυτές υποστηρίχθηκαν από την Προεδρία της χώρας, υποστηρίζονται επίσης και από διάφορες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δημιουργήσαμε επίσης και μια κεντρική υπηρεσία καταστολής του εμπορίου ναρκωτικών και ενισχύσαμε τον μηχανισμό καταστολής αυτών των δραστηριοτήτων. Σύμφωνα λοιπόν με τους στρατηγικούς άξονες του προγράμματος καταπολέμησης της ανασφάλειας και της τρομοκρατίας, Έχουμε κάνει τώρα ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα με μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας βαχυπρόθεσμα στον φορά της χώρας για την περίοδο 2010-2012. Βασικός στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να μειώσουμε με σημαντικό τρόπο ή και να καταργήσουμε εντελώς τις αιτίες ανασφάλειας στο Βόρειο Μαλί στα πλαίσια συγκεκριμένων ενεργειών, σοβαρών δράσεων και στα πλαίσια της ανάπτυξης των κοινοτικών δυνατοτήτων. Η στρατηγική αυτή ασκείται φυσικά από την δημόσια διοίκηση με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Ε, προσπαθούμε και σε επίπεδο διόρθωσης εκ των υστέρων αλλά και πρόληψης Προσπαθούμε να βελτιώσουμε επίσης και τις υποδομές τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιούν και στις οποίες πρέπει να βασίζονται οι αρχές ασφαλείας και οι στρατιωτικές αρχές για την καταπολέμηση του θρησκευτικού φανατισμού και της τρομοκρατίας γενικότερα. Η κυβέρνηση του Μαλή φυσικά και αναλαμβάνει ε, την κάλυψη των εξόδων των οικονομικών σχετικά με τους εξοπλισμούς και τις δαπάνες ε, που θα προκληθούν από τα προγράμματα αυτά. Θα δημιουργηθεί επίσης και μια επιτούτου συγκεκριμένη δομή ε, η οποία θα ανήκει στην κρατική διοίκηση αλλά θα επιτρέψει τον σωστό συντονισμό των διαφορετικών Υπουργείων που συμμετέχουν σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Κυρίες και κύριοι, το θέμα της περιοχής αυτής της υποσαχαρικής Αφρικής είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίσαμε στα πλαίσια μια σωστής ανάλυσης της περιοχής και των προβλημάτων της και ε, φυσικά στα πλαίσια των προτάσεων που ήδη από το 2006 εγώ προσωπικά είχα προτείνει, είχα προτείνει επίσης και μια διεθνή διάσκεψη για την ανάπτυξη και την ειρήνη στην υποσαχαρική αυτή ζώνη. Θα πρέπει να δεχτούμε λοιπόν να κατανείμουμε τις ευθύνε. Καμία από τις χώρες της ζώνης αυτής δεν μπορεί μόνη της να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και καμία από τις χώρες αυτές δεν είναι απαλλαγμένη από τις απειλές. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ την σοβαρή έλλειψη μιας υποπεριφερειακής μορφής συνεργασίας απέναντι σε προκλήσεις οι οποίες είναι διασυνοριακές. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας δεν αφορά την ασφάλεια μόνο, είδαμε ότι αυτό δεν αρκεί. Η καταπολέμηση της τρομοκρατίας αφορά την συμμετοχή των κοινοτήτων, των τοπικών αρχών, των τοπικών βουλευτών και της δημόσιας διοίκησης, αλλά σπονδυλική στήλη αυτής της προσπάθειας είναι η ανάπτυξη, η τοπική ανάπτυξη, έτσι ώστε να δώσουμε αναλλακτικέ δυνατότητες στις κοινότητες που κατοικούν στο βορρά του Μαλή. Η μαθητεία, η κατάρτιση μπορεί να βοηθήσει τις επιμελητιακές στην κάλυψη των επιμελητιακών αναγκών. Η καταπολέμηση των εγκληματικών δικτύων, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί συλλογικά από τις χώρες της υποσαχαρικής ζώνης. Έχω επιμείνει στην ανάγκη του να προσφέρουμε ένα νέο μέλλον στους κατοίκους της περιοχής αυτής. Θα ήθελα να προσθέσω ότι η κοινωνική πρόοδος και η ευημερία των πληθυσμών αυτών είναι κάτι το οποίο επιθυμεί το σύνολο των κατοίκων του Μαλή και γι' αυτό πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και εδώ τίθεται και το θέμα της επίτευξης των στόχων της χιλιετίας. Πήραμε κάποιες πρωτοβουλίες για την επιτάχυνση του προγράμματός μας. Πρόκειται για την πρωτοβουλία των 166 τοπικών αρχών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και στα πλαίσια λοιπόν των στόχων της χιλιετίας και στα πλαίσια των στόχων της αποκατάστασης της υγείας των κατοίκων της περιοχής. Γνωρίζουμε ότι όλοι οι στόχοι δεν θα στεφθούν από επιτυχία, δεν θα εκπληρωθούν, αλλά έχουμε κάνει βήματα προόδου και στον τομέα της πρόσβασης σε σχολεία και στον τομέα της πρόσληψης από τις πρόληψης του AIDS και στον τομέα της παροχής ποσίμου ύδατος. Ελπίζουμε λοιπόν ότι και η συνάντηση στη Νέα Υόρκη θα βοηθήσει έτσι ώστε να εφαρμοστούν σωστότερα τα προγράμματα τα οποία αφορούν την Αφρική, τι προσπάθειες θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω, πώς θα βελτιωθεί ο συντονισμός των προσπάθειών αυτών, πώς θα προλάβουν οι περιοχές οι οποίες σημειώνουν ειστέρηση χρονική και αυτό νομίζω ότι απαιτεί και τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθεια αυτή. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, κύριε εκπρόσωπε της ε, εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, ε, κυρίες και κύριοι, το Μαλί θα γιορτάσει σε δύο εβδομάδες τα 50 χρόνια ανεξαρτησίας. Θα ήθελα να μου επιτρέψετε να επιθυμίσω αυτό ότι η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την χώρα μας ε, τη στιγμή της ανεξαρτησίας της, δηλαδή στις 24 Σεπτεμβρίου του 1960. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε λοιπόν την Ευρωπαϊκή Ένωση για την σημαντική συμμετοχή της στην ανάπτυξη της χώρας. Η τιμή την οποία μου προσφέρετε σήμερα που με υποδέχεστε στην Ολομέλειά μας, Ολομέλειά σας μάλλον, μου δίνει ακόμα περισσότερες ελπίδες και πίστη στην προσπάθεια την οποία κάνουμε για να βελτιώσουμε τις σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας και φιλίας. Σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Uh, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζουμε τον πολιτικό διάλογο, όπως είπατε κι εσείς, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαλή. Μιλήσατε για τις μεταρρυθμίσεις στη χώρα σας. Οι μεταρρυθμίσεις είναι παντού αναγκαίες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπατε επίσης ε, για να υπάρξουν πολιτικοί συμβιβασμοί για ένα καλύτερο αφρικανικό μέλλον. Εμείς σας καλωσορίζουμε εδώ γιατί ακριβώς αυτό πράττουμε και εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα τελευταία χρόνια το ίδιο και εμείς προσπαθούμε να επιτύχουμε. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν ε, και ε, για την ομιλία σας σας ευχαριστούμε και για την παρουσία σας. Thank